Dear colleagues, αγαπητοί συνάδελφοι, νόμιζα ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. I Ξεκινώ με το σημείο 2 στην ημερήσια διάταξή μας που είναι η έγκριση της ιδίας αυτής της ημερησίας διάταξης. Έχω λάβει μια αίτηση τροποποίηση της ημερησίας διάταξης. Η ομάδα του ΕΛΚ έχει ζητήσει να αναβληθεί η ψηφοφορία για την έκθεση σε σχέση με το δικαίωμα στο νερό. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, Κύριε Μπόιλαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω, φαντάζομαι μάλλον ότι πολλοί απογοητεύονται από την ε, αίτηση για ε, για την ε, αναβολή αυτής της έκθεσης είναι μία από τις πρώτες εκθέσεις που έχουν να κάνουν με μία πρωτοβουλία πολιτών που είναι ένα σημαντικό δημοκρατικό δικαίωμα. Καταλαβαίνουμε τους τα προβλήματα της ομάδας του ΕΛΚ σε σχέση με τα χρονικά θέματα. Για μας είναι ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τη διαφάνεια. Γι' αυτό εμείς θέλουμε να ψηφιστεί η αίτηση ε, αναβολής με την οποία φυσικά διαφωνούμε. Ο Πέτερ Λίζε. Ευχαριστώ <clears throat> κύριε Πρόεδρε. κατανοώ την θέληση της ε, εισηγήτριας να ψηφίσουμε στο στον ταχύτερα, αλλά χρειάζεται κατανόηση στο γεγονός ότι εδώ έχουμε μια πρωτοβουλία πολιτών, Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, η πρώτη φορά που αντιμετωπίζεται στην Επιτροπή μας και μετά στην Ολομέλεια και εδώ ο κοινό μας ε, στόχος θα πρέπει να είναι να βρούμε ε, συμβαστικές λύσεις οι οποίες μπορούν να δοκιμήσουν στην Ολομέλεια. δεν είναι πολύ εύκολο να καταθέσουμε τροπολογίες στην Ολομέλεια. Γι' αυτό ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο να βρούμε συμβαστικές λύσεις στην ε, Επιτροπή μας. Εάν υπάρξουν νέα στοιχεία, φυσικά μπορεί να επανέλθει η συγγήτρια, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι θα λάβει χώρα. Μπορούμε λοιπόν να Θυμηθούμε ότι η έκθεση αυτή είχε αποδοθεί στην ΚΟΕ ήδη από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα που έλαβαν χώρα οι συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών, η δική μας εισηγήτρια, σκιώδης, είναι δυστυχώς ασθενής. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει μια αναβολή Εμεί ζητάμε τρει εβδομάδε. Εμεί πράγματι θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτή την έκθεση γιατί είναι όπως ελέγχθη η πρώτη φορά που έρχεται ω εδώ μια ε, πρωτοβουλία προ πολιτών, αλλά λόγω τη ασθένεια τη ε, σκιώδη εισηγήτριά μα δεν νομίζω ότι έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε για τι συμβαστικέ τροπολογίε γι' αυτό ζητούμε τρει εβδομάδε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ευρύτερε συμβαστικέ λύσει Θα ήταν κρίμα να περάσει μια τέτοια πρόταση με δύο μονάχα στην Επιτροπή μας και μετά να απορριφθεί στην ε, Ολομέλη. Αυτό δεν θα είναι θετικό ούτε και για την συγγητρία. Χρειαζόμαστε μια ευρία πλειοψηφία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όπως οφείλουμε στις αιτήσει των πολιτών. Γι' αυτό ζητώ αυτή την αναβολή κατά τρεις εβδομάδες. Η κυρία Γκαρσία Πέρεθ. Ευχαριστώ και εγώ καταλαβαίνω την σημασία που έχει η έκθεση αυτή. Έχω επίγνωση των δυσκολιών που έχουν ανακύψει στην ε, ομάδα του ΕΛΚ σε σχέση με την ε, διαδικασία διαπραγματεύσεων και εργαζόμαστε ήδη εδώ και δύο εβδομάδες προσπαθώντας να βρούμε συμβαστικές λύσεις αλλά αν πράγματι υπάρχει πολιτική θέληση στο σύνολο της Επιτροπής μας να φτάσουμε σε μια συμφωνία στην Ολομέλεια, πριν από την Ολομέλεια. Νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος περιμένει την ψηφοφορία από την Επιτροπή μας. Θα είναι ένα μήνυμα από την Επιτροπή μας προς την κοινή γνώμη για ένα σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται με την πρωτοβουλία πολιτών. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σήμερα την ψηφοφορία και με την κοινή βούληση όλων να βρούμε ένα τρόπο που συνάδει με τον κανονισμό ώστε να μπορέσει να γίνει μια συζήτηση στη συνέχεια, ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία εν ώψη της Ολομέλειας ή τουλάχιστον μια καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών ομάδων πριν από την Ολομέλεια. Okay. κανεί. Όχι. Πρέπει να ψηφίσουμε τότε. Α, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, λέει η κυρία Κονέτσνο. Θέλω να στηρίξω την εισηγήτρια. Ένα χρόνο έχει ξοδέψει δουλεύοντας πάνω σε αυτό το θέμα και πάρα πολλοί άνθρωποι, πολίτες, περιμένουν. Περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα, περιμένουν να δουν πώς και πότε θα εγκριθεί η έκθεση αυτή. Αν υπάρχει θέμα στο μέλλον, Πάντα κάποιος μπορεί να μην είναι παρόν, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να βοηθήσει. Δέκα μήνες έχουν περάσει που δουλεύουμε πάνω σε αυτή την έκθεση. Θέλουμε να προχωρήσει, έχουμε δουλέψει πάνω σε αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να δείξουμε σεβασμό σε όλους εκείνους οι οποίοι περιμένουν έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους δρόμους των ε, πολεών μας που περιμένουν να προχωρήσουμε με αυτή την πρωτοβουλία πρέπει να δείξουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι το κοινοβούλιο μας νοιάζεται και άρα να προχωρήσουμε. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην αναβάλουμε την ψηφοφορία. Δεν θα ήταν σωστό να ζητάμε την αναβολή τώρα μια-δυο ώρες πριν την ψηφοφορία. Θα έπρεπε να έχει συζητηθεί νωρίτερα αν υπήρχαν σοβαροί λόγοι. Αν το ΕΛΚΑ τα ήξερε, θα έπρεπε να το είχε πει νωρίτερα. Και όχι ήρθε στο βράδυ σήμερα το πρωί, τελευταία στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν Αγαπητοί συνάδελφοι, να στηρίξουμε την ψηφοφορία σήμερα και να ψηφίσουμε. Πρόεδρε, τα επιχειρήματα που ακούω είναι ότι την έκθεση αυτή πρέπει να την πάρουμε πολύ στα σοβαρά και συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Και ακριβώς επειδή η ομάδα μου, οι φιλελεύθεροι, οι άλλοι δεν πιστεύουν ότι είναι πολύ σοβαρή, γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να αναβληθεί η ψηφοφορία. Το τελευταίο που θα ήθελα να συμβεί είναι να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή εδώ στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και μετά να καταψηφιστεί στην Ολομέλεια. Τότε δεν βοηθάμε για αυτή την πρώτη πρωτοβουλία πολιτών. Αν λοιπόν την πρωτοβουλία πολιτών την παίρνουμε στα σοβαρά, πρέπει πραγματικά να αναβληθεί η ψηφοφορία. Τρει εβδομάδε καθυστέρηση δεν είναι τίποτα αν συγκρίνουμε με του μήνε που έχουμε περάσει δουλεύοντα πάνω στην πρωτοβουλία αυτή. Πρόεδρος, ωραία, ακούσαμε δύο υπέρ, δύο κατά, τώρα θα ψηφίσουμε. Παρακαλώ. Ίσως λέει κύριο κύριος Μπορώ να επανέλθω. Ο πρόεδρος διακόπτει. Είπα ότι κλείνει η συζήτηση. Έχω όμως άλλη πρόταση εγώ, διαδικαστικό. Δύο λεπτά να σταματήσουμε, ώστε οι συγγήτρια με τους σκιώδες να ε, μιλήσουν μεταξύ τους και μετά να αποφασίσουμε. Δύο λεπτά διακοπή. Προτείνω, λέει ο κύριος Γκρότε. If we want Πρόεδρος, εντάξει, αν θέλετε δύο λεπτά, ναι, αλλά μετά έτσι καλώς θα χρειαστεί να ψηφίσουμε ε, για το τι θα κάνουμε. Δύο λεπτά. Dear colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο Πρόεδρος, επιστρέψτε στις θέσεις σας παρακαλώ για να συνεχίσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Okay, we can Ωραία, τώρα αρχίζουμε. Πρέπει να ψηφίσουμε επί του αιτήματο αναβολής της ψηφοφορίας όσον αφορά το δικαίωμα στο νερό. Ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Ναι, ψηφίζει όποιος θέλει να αναπληθεί είναι υπέρ τη αναβολής, ρωτάει κάποιο. Όποιος είναι υπέρ τη αναβολής ψηφίζει ναι. Και κατά, όχι. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Everybody had voted. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα είναι ότι πρέπει να ψηφίσουμε κατά της αναβολής. Ψηφίζουμε λοιπόν. Αρχίζουμε λοιπόν και περνάμε στην ψηφοφορία για novel food. Πρώτα, συμφωνία με το Συμβούλιο. Ψηφίζουμε. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά για τα novel foods, νέα τρόφιμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις φοφορίες ναι. Εγκρίθηκε. Καζίνες τώρα. Μία ψηφοφορία έχουμε και εδώ να κάνουμε. Πρώτη ανάγνωση, συμφωνία με το Συμβούλιο για τις καζίνες. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά. Έχω έναν από τους πράσινους παραπάνω. Ωραία, ψηφίσατε όλοι πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. So, simple battle is finished. <laughs> complicated one on. Τώρα περνάμε στα πιο περίπλοκα για το νερό. Ναι. Κύριε Μπόιλα. Έχουν ζητηθεί ονομαστικέ ψηφοφορίε για τι συμβιβαστικέ. Ναι, όντω έχει ζητηθεί ονομαστική ψηφοφορία. Πρώτα εγκρίνουμε τις ονομαστικές ψηφοφορίες και νομίζω ότι είναι απλούστερο να γίνει ηλεκτρονικά αυτό. Ποιοι είναι υπέρ των ονομαστικών ψηφοφοριών, ψηφίζει ναι, οι άλλοι ψηφίζουν όχι, κατά. Ψηφίστε παρακαλώ. Has everybody voted? Ψηφίσατε όλοι. Ψηφίσατε όλοι. Πρόεδρε, κάποιος από την αίθουσα. Πέρασε. Πρώτη συμβιβαστική αριθμός 1. Με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 31. Σαβίνη. Υπέρ παρακαλώ. Διανατάσσεως της χειρός, ε. Δεν βλέπω όμως κανένα χέρι. Κατά. Απορρίπτεται. αποχές. Απορρίπτεται. ΔΕΒΕ 1 6. α 6 υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Θέλετε να ελέγξουμε την 5-6-β. Αναφορά 6. Ψηφίστε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. Ναι, αν δεν σηκώνετε τα χέρια, εντάξει, το αποτέλεσμα είναι προφανές, αλλά δεν έβλεπα χέρια. Τροπολογία 38, όχι, πέτη 8. Αναφερόν 8. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Γκαρσία. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Είναι η πρώτη φορά που κάνω ψηφοφορία. Παρακαλώ να είστε καλοί μαζί μου. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 36. Τέρμε. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχέ. Θα ελέγξουμε. Πέρα τη φοφορία. εγκρίθηκε. Τροπολογία αριθμός 1 αναφορών. 51α. Α, όχι, δεν την ψηφίζουμε. Συμβαστική 9 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Συνεχίζουμε με την τροπολογία 45. Τατσίνη. Υπέρ. Κατά. Απορρίφθηκε. Τέτη 17. Υπέρ. Κατά. Έγκρινατε. Τέτη 1 β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πέτη 5-3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα τη ψηφοφορίες. Όχι ακόμα. Τώρα. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 54. Λέει ο πρόεδρος. Α, συγγνώμη, λάθος. Συμβιβαστική 14 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της φοφορίας. Εγκρίθηκε. Τώρα περνάμε στην τροπολογία 54 Σαλβίνη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 55, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε δικαιωχά. Αυτή τη φορά. 57. Καπούτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59 έχει αποσυρθεί. Και περνάμε στην 62. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Πέρας της φοφορίες. Εγκρίθηκε. 60 υπέρ. 60. Κατά. Αποχές. Η ίδια πλειοψηφία 63. Όχι, όχι, καταπίπτει. 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 73 τώρα. Υπέρ. κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Πέρα στις οφορίας. Απορρίφθηκε. Πέτη 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 80. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 81. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 82. Με προφορική τροποποίηση. Υπάρχουν αντιρρήσεις στην προφορική, για την προφορική. Όχι. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 5η 12 β. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Α, να ελέγξουμε. Ωραία. Ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 16 με ονομαστική ψηφοφορία. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεβε 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική έξι μονομαστική ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 97. Γκαρσία Πέρες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας, εγκρίθηκε. Τροπολογία 100, υπέρ, κατά, Αποχές. Θα ελέγξουμε γιατί δεν βλέπω χέρια. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 101. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέτη 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πέτει 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 102 Γκέρλιν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 103 Τέρμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέτει 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 με ονομαστική ψηφοφορία μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Υπέρ 105. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται πετη 20α. Θέλετε να ελέγξουμε για την 106. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας. Πέτη 20α τώρα. Περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πέτη 22. Υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. 122. Καπούτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τι θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Συμβιβαστική 3 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. 127 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας, Εγκρίνεται. Τροπολογία 137. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Ας ελέγξουμε. Εντάξει. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρας της φοφορίας Εγκρίθηκε. 139. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 5 20β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίθηκε συμβιβαστική 7 με ονομαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. And what is close. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 5-4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε. Πέρας προφορίες. εγκρίνεται. Να σηκώνετε τα χέρια σας καμιά φορά, λέει ο πρόεδρος. Δεν είμαι καλός μάντης. 148. Φαρία υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 149 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε 150 υπέρ κατά αποχές έλεγχος Πέρα της ψηφοφορίες, Εγκρίθηκε. 151 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρα της ψηφοφορίες, Εγκρίνεται. Πέτει 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέτει 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καλά, ας ελέγξουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Με ναι, ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. ...162, α, συγγνώμη, συμβαστική 15 προηγουμένως. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 523 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 514 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 Curling υπέρ κατά αποχές απολύτω 173 υπέρ 173 διορθώνει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 171 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 169 όχι εκπίπτει. 174 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 175 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ εγκρίθηκε σας είπα εγκρίθηκε 175 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές <clears throat> έλεγχος για την 179 άρχεται πέρα στις οφορίες εγκρίνεται. 183 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προχωρούμε στην 521 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 524 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 525 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος, έλεγχος. Άρχεται. Πέρας φοφορίες. Εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 198 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται <clears throat> 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 201 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 203 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 205 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5.26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕ 18 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 ονομαστική κλίση άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 2.30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.32 καθώς και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. κατά αποχές εγκρινεται 233 υπέρ <clears throat> κατά αποχές απορρίπτεται. 2.34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.35 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Δεύε ΔΒ5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.41 <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 2.45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος για τη 2.45. Πέρας, εγκρίνεται. ΔΕΒΕ 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τεβε 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τεβε 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.46 υπέρ κατά αποχές έλεγχους Πέρας. Εγκρίνεται. 2.47 με προφορική τροποποίηση. Αντιρρήσεις. Όχι. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ Δεν ψηφίζουμε το τμήμα διαφόσον δεν ευδοκίμησε το πρώτο τμήμα. 2.48 με προφορική τροποποίηση. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.49 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.51 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9.4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε σε θεολογικές αναφορές. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά αποχές γκριν. Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε B <clears throat> υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύε C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒΔ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒΗ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒΓ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒH υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒI υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΔΒJ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. DVL υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ κατά αποχές έλεγχος. Πέρας. Απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για 17. Πέρας. Εγκρίνεται. 13 κατά αποχές. Ε, πρέπει να έχει εκπέσει βέβαια. Εκπίπτει διότι έχει γίνει δεκτή 17. Δεκαεννέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Όχι, δεν θέλει κανείς το λόγο. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην κυρία Μπόιλαν. If you want to leave, please speed up. Παρακαλώ, όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, σε επιταχύνουν για να μπορέσουμε οι υπόλοιποι να προχωρήσουμε. colleagues, we will we, we have to continue with, with agenda. So please. Συνάδελφοι, πρέπει να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Παρά λοιπόν τα πηγαδάκια, ε, θα συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψεων για τι ε, τροπολογίες ε, και όσον αφορά την μείωση των εκπομπών ρήπων από τα οχήματα. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Άλμπερτ Ντες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι. Έχω αναλάβει από τον κύριο αυτή την έκθεση και θέλω να πω τα εξή. Πιστεύω ότι καταρχήν οι περαιτέρω εργασίες μας για τις εκπομπέ από ελαφρά οχήματα και από μικρά εμπορικά οχήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Χωρίς την κατάλληλη απόφαση για το FDA δεν μπορούμε να σκεφτούμε για περαιτέρω όρια για τις εκπομπές οξυδίων του αζότου και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια πιο σταθερή βάση για καθαρότερες εκπομπές. Μόνο με το RDE θα έχουμε, την... θα έχουμε μια βάση για λήψη αποφάσεως. Αυτό θα μπορούμε να το έχουμε το Σεπτέμβριο. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις διάφορες πτυχές και το γεγονός ότι διευρύνεται και η σφαίρα εφαρμογής θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή οι εκπομπές μεθανίου φαίνεται ότι είναι πέραν των ορίων που προβλέπονται στην αντίστοιχη οδηγία. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία ανάγκη για να υπάρξει περαιτέρω περιορισμός. Η Κομισιόν θα πρέπει να επιφορτιστεί να διευκολύνει την ε, προσαρμογή της οριακής τιμής για το μεθάνιο. Αυτό μπορεί να γίνει μονάχα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας συναπόφασης. Μετά από συζήτηση με τους σκιώδεις εισηγητές έχω πάρει την υποστήριξή τους. Μια συγκεκριμένη πρόταση της Κομισιόν επομένω θα ήταν απαραίτητη, αλλά δεν υπάρχει καμία τέτοια ε, πρόταση. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και στον κανονισμό για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος να λάβουμε υπόψη και τις εκπομπές μεθανίου για να μπορέσουμε να κλείσουμε το κενό αυτό σε εθνιστικό επίπεδο και να αποφύγουμε τις, από, εκπομπές μεθανίου που πλήττουν το περιβάλλον. Η συμπερίληψη του μεθανίου στην οδηγία για το διοξίδιο του άνθρακος θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε ό,τι αφορά την επίτευξη των στόχων του 2020 είναι απαραίτητο να δημιουργήσουμε και μια ασφάλεια προγραμματισμού για την βιομηχανία ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων. Λαμβάνοντας υπόψη και τις τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν για την ε, μετασκευή των οχημάτων για να συμμορφωθούν με τους στόχους αυτούς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον κανονισμό 115 Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οριακές τιμές που βρίσκονται εκεί. Για την μετασκευή λοιπόν των οχημάτων θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι τρόποι, κάτι το οποίο είναι <clears throat> εφικτό ακόμα και αν δεν είναι επιθυμητό. Γι' αυτό η διαγραφή της παραγράφου για το μεθάνιο και η προσαρμογή στην ε, διατύπωση για το διοξείδιο του άνθρακος είναι ε, και θα πρέπει να συμπεριληφθεί και το θέμα της εκπομπής του μεθανίου στις περαιτέρω προσπάθειες για μείωση των ε, εκπομπών μετά το 2020. Πρέπει αυτό να τεθεί λοιπόν και στο θεματολόγιο της Κομισιόν. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της ε, σήμανσης της ε, βενζίνης, νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε περαιτέρω ε, πρόοδο. Δεν θα υπάρξει κανένα τεχνικό πρόβλημα για την βιομηχανία να προχωρήσει στην αντίστοιχη σήμανση. Είμαι έτοιμος για συμβαστικές λύσεις και είμαι έτοιμος να ακούσω την άποψη των συναδέλφων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την διεύρυνση του, της σφαίρας εφαρμογής σε οχήματα μέχρι 7,5 τόνων. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να επιβληθεί ένα τέτοιο βάρος στην βιομηχανία οχημάτων, αλλά είμαι έτοιμος να ακούσω τις απόψεις και των άλλων συναδέλφων. Χθες μίλησα με τον πρόεδρο Τζοβάνι Λαβία, λέγοντας ότι πρέπει να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τον Σεπτέμβριο. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει ακόμα να συζητήσουμε και είναι εξόχως τεχνικό το θέμα. Και δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε βεβαιασμένα και να πρέπει να καταλήξουμε σε συμβαστικές λύσεις με βεβαιασμένο τρόπο. Νομίζω ότι το Σεπτέμβριο θα έχουμε περισσότερες ε, γνώσεις για την πρόθεση της Κομισιόν σε σχέση με το ΑΔΕ. Γι' αυτό θέλω να ζητήσω την υποστήριξή σας. Δεν χάνουμε χρόνο με τον τρόπο αυτό αν ψηφίσουμε τον Σεπτέμβριο και μετά θα μπορέσει ακόμα μέσα στο 2015 αυτό το θέμα θα στο Ευχαριστώ. Thanks to reporter. Now round four. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ακούσουμε τους κοιόδης. Μάριαν Ντάλι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω αντιδρώντα σε ορισμένα πράγματα που είπε ο εισηγητή. Είναι πολύ θετικό που ακούσαμε ότι ο εισηγητή λέει πω είναι πρόθυμο να συμβιβαστεί για κάποια θέματα Δυστυχώς εγώ δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία του όταν μιλάμε για τις, ε, εκδοχέ, ε, τις ε, εκπομπές από τα οχήματα και ότι θα εφαρμοστεί αυτό από το Σεπτέμβριο. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, δεν έχουμε καμία εγγύηση ότι αυτό θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο. Έχουμε όμως κάτι με το οποίο μπορούμε να σημάνουμε τη διαφορά, αλλά όπου θα καταλέξουμε να το αναβάλουμε. Αν υπήρχε μια εγγύηση ότι αυτές οι εκπομπές ε, θα ήταν εγγυημένες από το Σεπτέμβριο, θα ήταν άλλο πράγμα. Έχω την εντύπωση ότι θα αναβληθεί για τόσο καιρό, ώστε να καταλήξουμε να κάνουμε κάτι αντιφατικό σε σχέση με αυτό που θέλαμε να κάνουμε καταρχήν. Και αυτό είναι μια ανησυχία που ήθελα να μοιραστώ μαζί σας γιατί εφόσον δεν υπάρχει εγγύηση, ε, δεν, δεν, είμαι βέβαια για το τι θα συμβεί. Ε, υπάρχουν εξή σημεία στα οποία θα ήθελα να εστιάσω ε, σήμερα. Θα ξεκινήσω ε, Το μεθάνιο, από το μεθάνιο που είναι γνωστό ως αέριο του θερμοκηπίου και δεν θα πρέπει να το εξετάσουμε μόνο στο πλαίσιο των ε, οδηγών των ε, αυτοκινήτων θα πρέπει να το περιορίσουμε ωστόσο ώστε να αποφύγουμε απεριόριστη εκπομπή αυτού του αερίου του, ε, θερμοκήπιου. Ε, το μεθάνιο θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνεται και ως ισοδύναμο του διοξιδίου του άνθρακα και στις δικές μας ε, τροπολογίες προτείνουμε αυτό το μεθάνιο να μετατραπεί σε, διοξίδι, σε, κουμπές διοξιδίου του άνθρακα. Όμως πριν από αυτό θα πρέπει να γίνει μια λεπτομερής ε, αξιολόγηση επιπτώσεων ώστε να αξιολογηθεί η, δυνατότητα πραγματοποίησης αυτής, αυτού του εγχειρήματο. Ε, για όλα τα στοιχεία θα πρέπει να γίνουν λεπτομερείς μελέτες αντικτύπου, για να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε τις απαιτήσει του κανονισμού. Θα χρειαζόταν δηλαδή μια φυσιολογική ε, νομοθετική διαδικασία. Τώρα, χωριστές ε, εκπομπές διοξιδίου και μονοξιδίου του ε, αζότου. Εδώ χρειάζεται να γίνουν περιορισμοί ώστε να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε πλήρως προς τις απαιτήσεις. Το να ορίσουμε μια συγκεκριμένη αξία για το διοξίδιο του αζότου θα βοηθούσε σε αυτή την ιδέα. Αυτή είναι η θέση που έχουμε με, μαζί με, και από την οποία προωθούμε με τις απολογίες μας, επίσης τονίζουμε την ανάγκη για εξελόγηση αντικτύπου. Για να δούμε ποιο θα είναι το έφολο, όφελος συγκεκριμένων όριων. Τώρα, όρια εκπομπών σε χαμηλές ε, σε χαμηλές θερμοκρασίες για το σιδρογονάνθρακα και για το μονοξίδιο του, του... άνθρακα δεν ε, υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Συμφωνούμε με την ε, πρόταση της ε, Κομισιόν, αλλά θέλουμε συναπόφαση και να γίνει και πάλι αξιολόγηση αντικτύπου για το για όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό το μέτρο. Τώρα, έχουμε το ανώτατο όριο το οποίο αναφέρθηκε και από τον εισηγητή. Εμείς στηρίζουμε τη μείωση του υπερβολικού και μη απαραίτητου βάρους για τις ε, επιχειρήσεις. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε πλατφόρμες που θα μπορούσαν να καλύπτουν ε, τις νομοθεσίες ε, τόσο ελαφρών οχημάτων όσο και των βαρέων οχημάτων. Αλλά σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε την πρόταση της Κομισιόν να αυξηθεί στα 5.000, 5.000 τόνους 5.000 ε, ε, κιλά ε, το ανώτατο όριο. Σημείο 5. Η εισαγωγή των μετρητών κατανάλωσης καυσίμων καθώς και των δικτών εκπομπών στα ελαφρά οχήματα. έχουμε έλλειψη συνειδητοποίησης των οδηγών, ιδιαίτερα στα συγκεκριμένα οχήματα που συζητάμε εδώ, ενώ ε, με τους μετρητές θα μπορούσαμε να έχουμε πιο συγκεκριμένη συμπεριφορά από πλευρά των οδηγών. Η Κομισιόν λέει 2-3% μπορεί να μειωθεί η κατανάλωση καυσίμων εάν αυτά τα δύο στοιχεία εφαρμοστούν ε, από κοινού στα ελαφριά οχήματα. Ωστόσο, Ακόμα και η συντηρητική εκτίμηση οδηγεί στην 1% εξοικονόμηση καυσίμων. Πιστεύουμε λοιπόν πως η διάταξη αυτή προσθέτει αξία στην ε, πρόταση. Τώρα, το τελευταίο μου σημείο είναι ότι θα πρέπει να σχεδιαστούν οι έλεγχοι ε, των εκπομπών με βάση πραγματικές συνθήκες οδήγησης έτσι ώστε να αντικατοπτρίζονται στις νομοθεσίες οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές, όπου οι εκπομπές είναι πιο, πιο ε, ψηλές. Κύριος Ντόρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο με την σύσταση αυτή. Θέλουμε και χαμηλότερο διοικητικό άχθος για τους παραγωγούς. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το σχέδιο αυτό έκθεσης και κάποιες τροπολογίες που στηρίζουμε προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στους παραγωγούς, στους κατασκευαστές δηλαδή οχημάτων. Και είναι καλύτερα να υπάρχει μία μόνο άδεια και να έχουμε τους 7,5 τόνους το βασικό είναι να έχουμε ευελιξία η οποία θα επιτρέπει και στους κατασκευαστές να εκφραστούν. Έτσι θα αποφύγουμε μονάδες παραγωγής οι οποίες θα κοστίζουν πιο πολύ. Πιστεύουμε ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαδικασίας συναπόφασης πάντως και όχι να έχουμε κατεξουσιοδότηση πράξης. Είμαστε υπέρ του να περιορίσουμε την αρμοδιότητα αυτή των κατεξοδότηση πράξεων. Να μειώσουμε δηλαδή τις αρμοδιότητες που έχουμε δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρέπει να σκεφτούμε και τις συνέπειες που θα έχει η παρουσίαση του μεθανίου, κατά πόσο δηλαδή το βάζουμε στα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να δημιουργεί δυσκολίες για οχήματα που έχουν πιο φυσικά καύσιμα. Ίσως πρέπει να προσπαθήσουμε να μειώσουμε και τις εκπομπές αυτές. Επίσης, στηρίζουμε τις τροπολογίες εκείνες οι οποίες προβλέπουν να μην έχει, όπως είπα και πριν, κατεξοδότηση πράξης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα και να λάβουμε υπόψη μας και το διοξίδιο του αζότου σαν εκπομπή. Κάτι άλλο που συζητάμε είναι μια τροπολογία για την χρήση των κινητήρων υδρογόνου και την εισαγωγή μιας ένδειξης κάθε φορά που γίνεται αλλαγή ταχύτητας, αυτό να φαίνεται σε κάποιο μετρητή. Αυτό θα μπορούσε να προσφέρει πλεονεκτήματα. Τέτοιοι κινητήρες μπορούν να είναι πλεονέκτημα χωρίς να έχουμε επιπλέον κόστος. Βέβαια, αναρωτιόμαστε για τα οικολογικά πλεονεκτήματα που μπορεί να ε, προσφέρει αυτό το σύστημα, αν το συγκρίνουμε με τις επιπλέον δυσκολίες που αναλαμβάνουν οι κατασκευαστές. Για τις δοκιμές πρέπει να το ξαναδούμε, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το Σεπτέμβριο. Τότε νομίζω μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη νομοθεσία η οποία να χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια. Ελπίζω να έχουμε τις ενδείξεις που χρειαζόμαστε το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι που ζητάμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση θέλουμε να δουλέψουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Μάσινερ εκ μέρους των φιλελεύθερων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εξ του Νίλ Στόρβαλτ, του σκιώτη μας εισηγητή, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι παρόν σήμερα πρώτα να διαβάσω το ποίημα μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους αδυσχεωρούς εισηγητές για την πολύ καλή συνεργασία. Το θέμα των εκπομπών από οχήματα έχει συζητηθεί στην Επιτροπή μας και έχουν κατατεθεί 120 τροπολογίες. Γενικά εμείς χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή και εκτιμούμε ιδιαίτερα τα θετικά στοιχεία. Η ρήπανση της ατμόσφαιρας είναι ένα σοβαρό πρόβλημα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αντιμετωπίσουμε. Τα οχήματα παίζουν μεγάλη σημασία ιδίω σε αστικέ περιοχέ για την ποιότητα τη ατμόσφαιρα και έχουν ένα σημαντικό ρόλο. Η τεχνολογία πηγαίνει προ τα εμπρό με μεγάλα και γοργά βήματα και δεν πρέπει εμεί να υπολοιπόμεθα αυτή. Συγχρόνω όμω θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη αντιμετώπιση ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ισοδίκαια αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και να μην καταλήξουμε σε πολιτικές οι οποίες αντιβαίνουν με τους στόχους μας αυτά που μας ανησυχούν περισσότερο, όπως και άλλες ομάδες, είναι η συμπερίληψη των κατεξουσιοδότηση πράξεων για ζητήματα που θεωρούμε ότι είναι κεντρικά για την πρόταση, όπως τα ισοδύναμα διοξιδίου του άνθρακος, τα όρια στο διοξίδιο του αζότου. Όλα αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι μόνο τεχνικά θέματα. αντίθετα θα λαμβάνουμε μια πλήρη έκθεση αντικτύπου και να έχουμε πλήρη πληροφορία για την εφαρμογή μια τέτοια απόφαση, προτού δώσουμε μια λευκή κάρτα, carte blanche στα ελληνικά, στην Κομισιόν. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν ήδη όρια για τα οξύδια του αζότου και εφόσον το διοξίδιο του άνθρακος είναι ένα από τα οξύδια αυτά, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να έχουμε μονάχα όρια για το διοξίδιο του αζότου. Αλλά μπορούμε να το συζητήσουμε. Ο στόχος αυτής της πρότασης είναι να μειωθεί η ρήπανση από οχήματα και θα πρέπει να επιτύχουμε το στόχο αυτό. Πιστεύουμε ότι μια δημοκρατική διαδικασία μέσω της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας είναι η καταλληλότερη και συγχρόνως δεν θα μειώσει το επίπεδο φιλοδοξίας μας. Υπάρχει λοιπόν καλό και έφορο έδαφος για συζήτηση για τα θέματα αυτά και θέλω να προσθέσω και το εξή, πέραν αυτό που είπε ο κύριος Τόρβαλτς, ότι συμφωνώ γενικά η Άλντε συμφωνεί ότι θα πρέπει να αναβάλουμε την εξέταση έκθεση αυτής μέχρι ότι η Κομισιόν μας ε, φέρει τα νέα στοιχεία για το RDA, δηλαδή για την δοκιμασία σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Επίσης, σε ό,τι αφορά την ε, ε, μέτρηση κατανάλωσης καυσίμων, τα περισσότερα αυτοκίνητα έχουν ήδη τέτοιους μετρητές και ακολουθώ αυτό το οποίο είπε η Επιτροπή Μεταφορών, όπου η πλειοψηφία ζήτησε να το κάνουμε αυτό σε εθελοντικό επίπεδο και να το αφήσουμε σαν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους κατασκευαστές που θέλουν να το εφαρμόσουν, επομένως δεν πρέπει να υπάρξει υποχρεωτική επιβολή. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω από την ΚΟΕ κάποιον σκιώδη από τους πράσινους. Ο Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πράγματι, την Κιφ Τέιλορ αντικαθιστώ. Δεν μπορούσα να είναι εδώ σήμερα δυστυχώς. Όμως θα μεταφέρω. Όπως και ζήν θα πω αναμειγμένα διάφορα στοιχεία. Συμφωνούμε βέβαια. Κοιτάξτε, συγκεκριτή γνωρίζει πάρα πολύ καλά, το έχει πει ότι είμαστε πολύ επικριτικοί πάνω στην πρόταση αυτή. Πρώτα απ' όλα, ο τίτλο είναι Μείωση των ρηπογόνων από το χήματα Εμεί δεν έχουμε την αίσθηση όμω με την έκθεση αυτή, όντω κάνουμε αυτό που λέει ο τίτλο γιατί εδώ βλέπουμε περισσότερη ευελιξία. Αυτό μόνο προτείνεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ίσως θα έπρεπε τουλάχιστον να αλλάξει τον τίτλο. Γιατί δεν πρόκειται για μείωση τελικά των ρηπογόνων καθάλλου. Εκτός βέβαια αν τροποποιήσουμε την έκθεση, οπότε τελικά η ρύθμιση αντικατοπτρίζει αυτό που ανακοινώνει ο τίτλος. Αλλιώς δεν μπορούμε να στηρίξουμε εμείς την πρόταση αυτή. Όπω το γνωρίζει και ο εισηγητή, είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί. Υπάρχουν δύο στοιχεία κλειδί για μα. που από αυτά θα εξαρτηθεί το κατά πώς θα στηρίξουμε ή όχι. Το πρώτο το έχει ξαναπεί ο Κιφ Τέιλορ. Κατά τη γνώμη μα, πρέπει οι απαιτήσει να είναι υποχρεωτικέ όσον αφορά του μετρητέ κατανάλωση καυσίμων και του δείκτες αλλαγή ταχύτητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα λέει ότι πρέπει να γίνονται εκθέσει αντικτύπου και πάντα λένε ότι για να έχουμε καλύτερη ρύθμιση η καλύτερη λύση είναι να έχουμε τέτοιες εκθέσεις αντικτύπου. Ε, λοιπόν, εδώ ότι έκπληξη δεν ακολουθεί τη δικιά της έκθεση αντικτύπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν άρεσε ίσως στην βιομηχανία, αλλά αυτός δεν είναι λόγος να μην τη συμπεριλάβουμε. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μειώσουμε τις εκπομπές. Το λέει η έκθεση αντικτύπου, γι' αυτό και εμεί θέλουμε να είναι υποχρεωτικοί οι μετρητές κατανάλωσης καυσίμων και δείκτες αλλαγής ταχύτητας. Αλλιώ δεν έχει νόημα αυτή η έκθεση και να τη αλλάξουμε τίτλο τουλάχιστον. Το δεύτερο που έχει ήδη αναφερθεί και εδώ στηρίζουμε τον εισηγητή να αναβληθεί η ψηφοφορία στην ΕΝΒΗ. Και αυτό έχει να κάνει με τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ακούγεται πολύ αθώο να αυξήσουμε τη μάζα ώστε και τα πιο βαρέα οχήματα να ανήκουν στην κατηγορία των ελαφρών, αλλά το θέμα είναι οι πραγματικές συνθήκες οδήγησης, οι δοκιμές δηλαδή σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Ξέρουμε ότι τα βαρέα δεν μπορούν να είναι στην κατηγορία των ελαφρών. Λοιπόν, όσο δεν καλυφθεί αυτό, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε για το εύρος εφαρμογής. Το εύρος εφαρμογής ακούγεται έτσι πάρα πολύ ωραίο τεχνικό θέμα, αλλά είναι πολιτικό τελικά. Πολύ πολιτικό. Γιατί αν δεν έχουμε εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες ε, οδήγησης για τα ελαφρά, δεν βλέπω πώς θα διευρύνουμε το εύρος εφαρμογής. Συνεπώς και εμείς και συμφωνούμε. Δεν ξέρω τελικά θα έχει γίνει το Σεπτέμβριο, αλλά όλα αυτά έχουν τόσο μεγάλη σχέση μεταξύ τους που είναι δύσκολο να πούμε ότι μπορούμε να τα χωρίσουμε. Πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε λοιπόν να γίνει η απόφαση για τις ε, δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης και μετά να προχωρήσουμε. Και αυτό για μας είναι στοιχείο κλειδί λοιπόν αυτά τα δύο. Μόνο τότε μπορούμε να προχωρήσουμε. Φυσικά υπάρχουν και άλλα που αναφέρθηκαν. Πολύ σύντομα θα σας αναφέρω όλα τρία. Πρώτον, Είμαστε κατά της εξαίρεσης ε, των εκπομπών ε, οχημάτων με φυσικό αέριο. Δεν βλέπουμε γιατί υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Οπότε δεν θα συμφωνήσουμε με την εξαίρεση αυτή. Είμαστε επικριτικοί και σε πολλές από τις τις πράξεις που προτείνονται, γιατί δεν είναι τεχνικά ζητήματα αυτά, είναι καθαρά πολιτικά. Σίγουρα όταν πρόκειται για το καθορισμό ορίων εκπομπών ρήπων. Οπότε εδώ νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε και με άλλους συναδέλφους. Και το τρίτο και τελευταίο, δεν στηρίζουμε ένα χωριστό όριο για το διοξίδιο του αζότου. Χρειαζόμαστε ένα γενικό όριο για όλα τα οξύδια του αζότου. Δεν έχει νόημα να βάζουμε χωριστά όρια για το διοξίδιο του αζότου. Και συμφωνούμε με το Κασίνη και με άλλους. Αυτά λοιπόν είναι τα τρία. Ναι, Ματίας, ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν αισθάνεσαι και πολύ καλά τώρα. Ε, κι εγώ άλλες φορές έχω βρεθεί σε αυτή τη θέση. Πάντως μην ανησυχείς, μια χαρά θα τα πάμε. Πάντως τα βασικά στοιχεία κλειδί είναι οι πραγματικέ συνθήκε εργασία όπω σα είπα και η υποχρέωση για μετρητές κατανάλωσης καυσίμων και δικτών αλλαγής ταχύτητα. Αυτά λένε ο Κίθ Τέλος και εγώ που έχω προσθέσει και εγώ μερικά σε αυτά του Κίθ. Ευχαριστώ πολύ για τα <clears throat> σχόλια σα. και τώρα η κυρία Ήβη για το EFTD. Σας ευχαριστώ. Και εμείς συμφωνούμε να συμπεριληφθεί το μεθάνιο ανάμεσα στα συστατικά των, ε, του συνόλου των εκπομπών υδρογων ανθράκων. Ε, θέλουμε να μείνει στη... Μπορούμε να συζητήσουμε τα όρια, αλλά όχι την αφαίρεση τους. Ε, ε, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την επιρροή του μεθανίου και των υποβαθμισμένων του προϊόντων στην ατμόσφαιρα για να έχουμε ένα συλλογικό περιβαλλοντικό μέτρο. Συμφωνούμε επιπλέον στο να ορίσουμε νέα όρια για το διοξίδιο του αζότου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία αυτού του συστατικού για την ανθρώπινη υγεία, πράγμα που φαίνεται και από το τελευταίο έγγραφο που δημοσίευσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για το Περιβάλλον για την ανθρώπινη υγεία. Ε, Έχουμε επίσης οι δοκιμές θα πρέπει να γίνονται υπό πραγματικές συνθήκες οδήγησης, όμως ε, δεν συμφωνούμε να γίνονται αυτές οι αλλαγές με κατεξοδότηση πράξη. Από τη στιγμή που ο, ορισμός, ε, που κανονισμός μάλλον αφορά συγκεκριμένα όρια εκπομπών, δεν μπορεί να θεωρείται ότι δεν είναι νομοθετικό κείμενο. Η μόνη λύση λοιπόν που είναι να παρουσιάσει η Κομισιόν ε, μια νέα πρόταση που θα συνοδεύεται από μελέτες αντικτύπου τύπου και θα εξεταστεί σύμφωνα με την ε, συνηθισμένη διαδικασία συν απόφαση. Σας ευχαριστώ πολύ. Άλλοι συνάδελφοι τώρα. Ματίας. Ευχαριστώ. Το Ευρώ 5 και το Ευρώ 6 ξεκίνησαν αυτές τις διαδικασίες πριν από 10 χρόνια σχεδόν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους ότι τότε είχαμε εισαγάγει μια ειδική ε, σειρά διατάξεων για τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν σχέση με κοινωνικές παροχές. Και γι' αυτό έχω κάνει αυτή την ε, παράκληση προς τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές ώστε να μπορέσει να ακολουθηθεί αυτό και στη νέα νομοθεσία. Για μένα θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την εξαίρεση για αυτά τα οχήματα. Σε σχέση με τον κύκλο δοκιμασίας οχημάτων, δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε ακόμα περισσότερο στον ε, κατασκευαστή. Όλο και περισσότερα γκάτζετς έχουν τα αυτοκίνητα Επιτρέπεται βέβαια στις δοκιμασίες να κάνουν διάφορα κόλπα οι καταναλωτές με αυτά τα gadgets. Είναι απαραίτητο να καθορίσουμε σαφώς τον ε, κύκλο δοκιμασία των αυτοκινήτων. Δεν θέλω όμως αυτό να καθυστερήσει 10 χρόνια αυτό το νομοθέτημα. Θα ήθελα το Σεπτέμβριο να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και ελπίζω ότι θα είναι ο Σεπτέμβριο του 2015 και όχι ο Σεπτέμβριο του 2016 ή ο Σεπτέμβριο του 2022. σχόλιο του κύριου χωρίς ε, ε, μικρόφωνο, μάλλον αναφέρεται στο αεροδρόμιο του Βερολίνου. Νομίζω ότι τελικά θα πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη αυτήν προσαρμογή, η οποία θα πρέπει να έχει συνεκτικό χαρακτήρα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη γραμμή που έχουμε ακολουθήσει τα τελευταία δέκα χρόνια και αν μπορεί να υπάρξει αυτή η εξαίρεση για τα κοινωνικού χαρακτήρα οχήματα. Θα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Είναι ένα μικρό τομέα οχημάτων, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τι μικρέ και μεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα, λέει ο κύριο Γκρότε. Κυρία Λουκαυσεύσκα, που είναι σκιώδη, είναι συντάξη τη ΤΡΑΝ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει το θέμα αυτό ήδη και στην Επιτροπή Μεταφορών. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο, ξέρουμε ότι είναι εξόχως τεχνικό το θέμα αυτό και έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε με τους εμπειρογνώμονες της Κομισιόν και με τους ενδιαφερομένους τους εκπροσώπους των κατασκευαστών. Ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε μέχρι ποιου βαθμού η πρόταση της Κομισιόν θα έχει επιρροή στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, αλλά συγχρόνως θα επηρεάσει και την αγορά των ε, ιδιωτικών οχημάτων, αλλά και των ελαφρών εμπορικών οχημάτων ξέρουμε ότι η ρήπανση της ατμόσφαιρας της πόλης είναι αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό των ε, οχημάτων. Ιδίως των ελαφρών οχημάτων. Ξέρουμε λοιπόν ότι τα οχήματα diesel είναι αυτά τα οποία ρηπαίνουν περισσότερο πια. Πριν από μερικά χρόνια θεωρούσαμε ακόμα ότι τα δίζελ ήταν τα καλύτερα και ήταν τα πιο κατάλληλα για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Αλλά τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι. Έχουμε την πρόταση της Κομισιόν. Το ερώτημα είναι τώρα αν πρέπει να είναι η βενζίνη ή το φυσικό αέριο ή αν θα πρέπει να δημιουργήσουμε περισσότερες, ε, περισσότερα κίνητρα για οχήματα τα οποία εκπέμπουν πολύ λιγότερους ρήπους. Έχουμε λοιπόν συζητήσει όλα αυτά τα θέματα με τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Υπάρχουν πολλά αμφίμαχα θέματα, υπάρχουν ε, κάποιες αμφιβολίες και επιφυλάξεις ιδίως με το ανώτατο όριο για, τα, για τις εκπομπές του άνθρακος. Υπάρχουν επίσης επιφυλάξεις σε σχέση με τη δημιουργία εισοδημάτων, ε, ισοδυνάμων για τα, το διοξείδιο του άνθρακος παραγωγικά για το μεθάνιο. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επωφελείς συμβιβαστικές λύσεις <clears throat> και ελπίζω ότι εδώ στην Επιτροπή ΕΝΒΗ θα μπορέσει να σας βοηθήσει η γνωμοδότησή μας. Οι στόχοι μας ήταν δύο. Πρώτα φυσικά να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, αλλά θα θέλαμε επιπλέον να δούμε ε, πώς θα επηρεάσει αυτό και την βιομηχανία και αν θα έχει ως αποτέλεσμα μια μείωση των θέσεων απασχόλησης. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσετε στην εργασία σας να επιτύχετε να αντιμετωπίσετε τα θέματα αυτά. δούμε λοιπόν τι θα βγει. Next speaker, Mr. Dems. Thank you, Chair. Um, I, I wanted to speak because obviously this is a source level piece of Ήθελα να μιλήσω γιατί πρόκειται για μια σημαντική ε, ε, νομοθεσία και εργάζομαι ως ε, εισηγητής και για την οδηγία για τις εθνικές εκπομπές και νομίζω πως αν η, νομοθεσία πηγή δεν είναι επαρκώς στεναρή, δεν θα μπορέσουν οι χώρες να την εφαρμόσουν. Θέλω λοιπόν να επανέλθω στα σχόλια της κυρίας Ντάλη. Όσον αφορά την εξασφάλιση ε, του ότι θα έχουμε σωστά τα στάνταρ ε, της πραγματικής οδήγησης, ε, ε, και ξέρουμε βέβαια ότι πρόκειται 22 φορές παραπάνω από την νόμιμα αποδεκτή ποσότητα για το μονοξίδιο του αζότου, ας πούμε, σε πραγματικές συνθήκες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να ε, το πετύχουμε, να το κάνουμε σωστά. Φοβούμε λοιπόν πως αν δεν γίνει αυτό ε, δεν θα λύσουμε κάτι ε, από όλα αυτά τα προβλήματα. Πρέπει πραγματικά να έχουμε συνθήκες πραγματικής οδήγησης ε, στους κύκλους δοκιμών όσο γίνεται πιο σύντομα. Δεν μπορούμε όμω αυτό να το αφήσουμε στου άλλου. Εμεί πρέπει να πιέσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνει. Και νομίζω πω είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη την τα αυτοκίνητα, τους κινητήρες μάλλον πετρελαίου εντός αστικών κέντρων όταν έχουν ε, όταν δηλαδή λειτουργούν ε, συνέχεια σταμάτα ξεκίνα, σταμάτα ξεκίνα στα ποτηλιαρίσματα και είναι τελείως διαφορετικές οι εκπομπές. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να το σκεφτούν πολύ προσεκτικά. Επίσης θα ήθελα να υποστηρίξω την ιδέα ότι έχουμε το μεθάνιο και ως ε, ρήπο ε, ε, στην ατμόσφαιρα αλλά και ως αέριο του θερμοκηπίου. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή νομοθεσία που να εξετάζει το μεθάνιο συγκεκριμένα ως αέριο του θερμοκηπίου και μάλιστα είναι αίτιο σοβαρών προβλημάτων υγείας εντός των πόλεων. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε μήπως πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένη στόχευση στο μεθάνιο. Ευχαριστώ. Και τώρα ευχαριστώ και η Κομισιόν να πάρει το λόγο τώρα για να απαντήσει στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους πήραν το λόγο και ιδιαίτερα τον εισηγητή και τους σκιώδης για τη δουλειά που έκανε. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα πολύ σημαντικό σχόλιο. Σε σχέση δηλαδή με τούτο εδώ το φάκελο και το φάκελο RDE που συζητιέται στην Επιτροπή. Είναι βέβαιο ότι οι κανόνες RDE είναι πολύ σημαντικοί για οποιοδήποτε φάκελο που ασχολείται με εκπομπές. Και βεβαίως πάντοτε θα υπάρχουν ε, δεσμοί με το αντί, Ωστόσο, η αναβολή μπορεί να προκαλέσει, όπως είπαν κάποιοι βουλευτές, ε, μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από αυτό που προσπαθεί να λύσει. Είναι αλήθεια ότι θα έχουμε κάποιες επιτυχές ε, ε, του RD, αλλά μόλις το Σεπτέμβριο. Αν γνωρίζετε ότι έχει υιοθετηθεί ε, πρόσφατα σε επίπεδο επιτροπής υπάρχουν διάφορα βήματα σε αυτή τη διαδικασία. Το Σεπτέμβριο θα γίνει ένα από αυτά τα βήματα. Θα έχουμε δηλαδή κάποιες οριακές τιμές, ελπίζω μέχρι το Σεπτέμβριο, ούτε και αυτό δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα τους ε, εγκρίνει τα όρια η επιτροπή του Σεπτέμβριου. Ελπίζουμε. Αλλά, ωστόσο, οι οριακές τιμές αυτές δεν θα, δεν θα ισχύσουν παρά μόνο στον επόμενο χρόνο ε, και δεν θα εφαρμοστούν πλήρως παρά μόνο μετά από κάποια χρόνια. Άρα λοιπόν ο αντίκτυπος των κανόνων RD ε, θα φανεί μετά από χρόνια. Θέλουμε λοιπόν να περιμένουμε ακόμα χρόνια μέχρι ότου να εγκρίνουμε τούτα εδώ τα όρια. Η Κομισιόν ελπίζει πως όχι. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα που θέλαμε να σας απευθύνουμε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Τώρα. Κύριε Ντες. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους, όλους τους κοιόδης εισηγητές. Νομίζω σε πολλά σημεία υπάρχει μια γενική συνένεση και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε αυτές τις συμβαστικές λύσεις οι οποίες μπορούν να περάσουν στη συνέχεια με μεγάλη πλειοψηφία. Δεν θα αντιδράσω τώρα σε όλα αυτά τα οποία ελέγχθηκαν. Θέλω να σταθώ σε μερικά <clears throat> βασικά στοιχεία εγώ. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα να, να βρούμε τρόπους να δώσουμε μια μεγάλη, μεγαλύτερη ασφάλεια στην ε, βιομηχανία, εάν κατέβουμε στα 90 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο διοξιδίου του άνθρακος, τότε θα πρέπει να, να αντιμετωπίσει η αυτοκινητοβιομηχανία αυτή την πρόκληση. Δεν μπορούμε από την πίσω πόρτα να εισαγάγουμε τέτοιες ρήτρε που θα εμποδίσουν την βιομηχανία να έχει ασφάλεια σχεδιασμού. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως και πολλοί που έλαβαν το λόγο χρειαζόμαστε μια καλύτερη αξιολόγηση από την πλευρά της Κομισιόν. Και επίσης οι οριακές ε, τιμές δεν μπορεί να αλλάζουν με κατεξουσιοδότηση πράξης. Παρά το γεγονός ότι οι κατεξουσιοδότηση πράξεις εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα του Κοινοβουλίου στο να βρίσκεται στη συναπόφαση, όπως είδα πρόσφατα στην Επιτροπή Γεωργίας. Πρέπει να διαπραγματευτεί μαζί μας η Κομισιόν για να προχωρήσει τα θέματα αυτά. Εμείς φυσικά πρέπει να διατηρήσουμε τα δικαιώματά μας ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρ' όλα αυτά έλω να διατηρηθούν οι τιμές οριακές ως αντικείμενο ε, συναπόφασης. Σε ό,τι αφορά τώρα την, ανα, την αναβολή, δεν είναι να το πάμε το Σεπτέμβριο και μετά Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο και τον επόμενο χρόνο, όπως άφησε να εννοηθεί ο κύριος ε, Κρότερ Εμείς δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα κατάλογο ψηφοφορίας χωρίς να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που να είναι όριμη η ψηφοφορία. Δεν μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε σε επίπεδο βεβαιασμένο για όλα αυτά τα θέματα. Πρέπει να υπάρξει σωστή διαχείριση του χρόνου ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε στις συμβαστικές μας προτάσεις. Χρειάζεται λοιπόν ένα χρονικό διάστημα από την ε, διατύπωση των τροπολογιών μέχρι την τελική ψηφοφορία. Γι' αυτό ε, επιμένω ότι πρέπει να έχουμε ψηφοφορία το Σεπτέμβριο και εφόσον δεν υπάρχει η πρόταση της Κομισιόν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα πριν από το Σεπτέμβριο. Και για τα ειδικά οχήματα κοινωνικού χαρακτήρα κύριε Κρότε θα πρέπει να βρούμε κάποια λύση. Δεν νομίζω ότι εδώ θα, δημιουργήσουμε, θα, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο παραθυράκι και ούτως ή άλλως όλα τα αρχήματα θα πρέπει να μειώσουν την ε, προστασία της ατμόσφαιρας, της από την ε, ρήπανση. Επίσης για το φυσικό αέριο οι Ρώσοι μας είπαν ότι υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται σταθμοί πεπιεσμένου φυσικού αερίου και αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα συνάδει και με τους στόχους της κλιματικής αλλαγής. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε ένα καλό δρόμο για να συμφωνήσουμε και να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λογικές ε, λύσεις και όπως είπα είμαι να ακούσω την άποψη των σκιωδών εισηγητών σε ό,τι αφορά τους δείκτες κατανάλωσης στα οχήματα. Εγώ πάντα κοιτάζω στο αυτοκίνητό μου τι καταναλώνω. Αλλά πολλές φορές υπάρχει μία διαφορά ανάμεσα στην, στην ενδείξεις και στην πραγματικότητα που μπορεί να ξεπεράσει το 2 ή 3%. Δεν υπάρχει φυσικά απόλυτη ακρίβεια, αλλά οι δείκτες κατανάλωσης τουλάχιστον δίνουν κάποια ένδειξη για το προς τα που κινείται η κατανάλωση υπάρχει ακόμα και σε οχήματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά. Μπορεί να υπάρξει φυσικά και το εθελοντικό, ε, η εθελοντική συμμόρφωση των αυτοκίνητων βιομηχανιών, αλλά εγώ νομίζω ότι η πλειοψηφία θέλει να υπάρξει υποχρεωτική παροχή πληροφοριών για την κατανάλωση. Λοιπόν, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Απλώς τονίζω ότι είναι πολύ πιο λογικό να ψηφίσουμε το Σεπτέμβριο. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστώ όλους για τη συζήτηση που είχαμε διάφορα τώρα. Δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Επόμενη συνεδρίαση 15 και 16 Ιουλίου στις Βρυξέλλες. Τελειώσαμε για σήμερα και σας ευχαριστώ.